morning to everybody. Dear we have to... Καλημέρα, συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε την, το σχέδιο γνωμοδότησης για τη μακροοικονομική ε, συνδρομή προς την Ουκρανία. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, η ημερήσια εγκρίνεται. Δεν έχω καμία αναγγελία του Πρόεδρου. Εάν έχετε σχόλια για τα πρακτικά, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Και ξαναλέω, ε, περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία Σχετική γνωμοδότηση. 27 ε, Σοφοζέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 Σοφοζέρ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 σόλτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. τέσσερα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Να προχωρήσουμε. 43 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 44 ε, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται, συγγνώμη και 43. 47 Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό για όλες. Όλες κυρία Πρόεδρε, όλες. 47 έως 54 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μπλοκ. 47 έως 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται όλες. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Α, ναι, εννέα. Υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Θέλετε να κάνω έλεγχο. Εγκρίθηκε, ωραία. 10. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10... 14 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ 16-19, 16-19 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. Μετά συμβαστική πρώτη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά 22-24, μπλοκ, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτονται. Μετά συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και την 4, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Εκοσιοκτώ 28 του κυρίου Κάρβερ. Την πηδήξαμε. Κύριε Κάρβερ, υπέρ, 28, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και 31 του κυρίου Σόλτς υπέρ, κατά, αποχές. Και πάλι, 31, 31, υπέρ, στην αρχή του καταλόγου, πρώτη σελίδα, 31, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και 35, και αυτή την ε, τη δείξαμε, ε, του κυρίου Κάρβερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα, ηλεκτρονική. της ψηφοφορίας Με συγχωρείτε, ο κύριος ε, Γκάλερ να πω ότι ζητά συγγνώμη για την απουσία του, αλλά θέλει να ενημερώσει για τις εξελίξεις ε, του φακέλου αυτού στην ΙΝΤΑ. Ο κύριος Βαλέσα επεδίωξε συμβαστική ε, με κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στο θέμα αυτό, οπότε ο κύριος Γκάλερ θα δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και πώς θα διαμορφωθεί το παρακολουθεί πάντω το θέμα, είναι στην επίσημη διαπραγμα... Ε, αντιπροσωπεία για την Νότια ε, Next one. Επόμενη ψηφοφορία. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο έκθεση ε, του κυρίου Νόριτσα Νίκολαε. Συστάσει προ το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΙΕΤ σχετικά με τι διαπραγματεύσει για τη Συνολική Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αζερβαϊτζάν. Για να είμαστε συνεπεί, θα ήθελα να σα θυμίσω ότι η δουλειά μα πάνω στην έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την έκθεση του κυρίου Ντόκε για την νέα Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία και το σχετικό ψήφισμα. Θα τα ψηφίσουμε αυτά αμέσως μετά την έκθεση για το Αζερβαϊτζάν. Ενημερώθηκε ο πρόεδρος ότι υπάρχουν 268 τροπολογίες. Ο μεγάλος αριθμός αυτών σχετίζεται με τη σύγκρουση των Αγκόρνο Καραμπάκ. Και πολλές ε, είναι ε, πανομοιότυπες. Θα ήθελα να σας, σας θυμίσω ότι η έκθεση αυτή αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν και η Επιτροπή μας δεν είναι απαραίτητα το κατάλληλο μέρο για να συζητάμε συνέχεια όλες τις πτυχές αυτής της σύγκρουση. Τέλο, ο Πρόεδρος ε, επικροτεί τι προσπάθειες για επίτευξη συμβιβασμών ε, αποδεκτών και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή το μήνυμα της έκθεσης αυτής θα πρέπει να σχετίζεται με τις προτεραιότητές μας ε, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Forty. Forty. Επαλήθευση της 40. Επαλήθευση της 40.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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 107, για να είμαστε βέβαιοι. Λήξη της ψηφοφορία.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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Όχι λάθος, προφορική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εύκολα τα πράγματα. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 259 του κυρίου Σόλς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. η Ηλεκτρονική επαλήθευση. Σόλτς. 259. I close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 υπέρ, 28 κατά. Δίκιο είχα. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Συμβαστική 31. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 της κυρίας Νικολάη υπέρ κατά κατά αποχές. Δεν είμαι βέβαιη. Ας το επαληθεύσουμε. I close the vote. πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 42. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αποσύρεται και μετά έχουμε την 35 υπέρ κατά αποχές σας παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 39. 39. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Αιτιολογικές αναφορές. 1, 2, 3 από κοινού. Υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ωραία. Δεν είμαι και βέβαιη. 8 και 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ζόφκο. 11. Υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 11. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γιατί δεν τα χέρια σας. 12 και 13 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση, 12 και 13. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 14, 15 και 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 17, 18, 19. Α, όχι, λάθος. 17, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Τις 17, παρακαλώ. Κανείς δεν σκόνει το χέρι του. Πέρα στις ψηφοφορίες, εγκρίνεται. 18 της κυρίας Γκόμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφής η κατάσταση. 19 παρακαλώ. 19. Nobody's raising hands. I close the vote. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές. 21. Θέλετε επαλήθευση της 21? Ωραία, πάμε πίσω πάλι. 21. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Καστάλτο Κοράο. Πέρασε ψηφοφορία για την 21. Απίστευτο, απίστευτο. Ευχαριστώ. Εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σας, θα αναγκαζόμαστε να επαληθεύουμε συνέχεια. 22 λόπε, υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, Αποχέ. η ηλεκτρονική επαλήθευση της 24. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και φτάνουμε τώρα στην τελική ψηφοφορία, η ηλεκτρονική. I close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην κυρία Νικολάη. Προχωράμε τώρα κατευθείαν στην συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια και των κρατών μελών του αφενό και τη Δημοκρατία τη Αρμενία αφετέρου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωράμε στο σημείο 7 νομίζω. Ψήφισμα που συνοδεύει την έγκριση για τη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια και των κρατών μελών του αφενό και τη Δημοκρατία τη Αρμενία αφετέρου. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15. Ναι, 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 17.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 Πέρα στις ψηφοφορίες. Αλλά πρέπει να σκόνετε τα χέρια σας. Εγκρίνετε. Παρακαλώ να συνεργαστείτε κι εσείς. Ε, συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73. Όχι, καταπίπτει. Ε, συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Η τροπολογία 73 καταπίπτει. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, προφορική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σόλς 90. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Μα τι να πω, αν δεν σκόνται τα χέρια σας, αναγκαζόμαστε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προχωράμε. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικέ σκέψει. 8. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές. 1. Τάνοκ. Υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα Πέρας της εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση. I close the vote. Πέρα στις ψυχοφορίες. Number three. Η τρία υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τέσσερα υπέρ. Τέσσερα και πέντε μαζί. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέσσερα και πέντε. I close the vote. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απίστευτο, απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθεση της 7. Παρακαλώ. adopted, such a bit close the vote. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος. Πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και προχωράμε στο σημείο Okay, don't worry. Don't worry. So... Άμυνα στον κυβερνό χώρο. Εισηγητής Ούρμα Σπάιτ. Ένα Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 138. Donjon. Τροπολογία Donjon 138. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 151. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154. Κάρβερ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 155. Υπέρ κατά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 Εγκρίνεται. 165. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 166. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 175. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 πάμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συγγνώμη, την 193, καταπίπτει. Απορρίπτεται. Εντάξει. Η 192 εγκρίνεται, η 193 καταπίπτει και η 194, 196 ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα της 196. 196 υπέρ το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 196. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν έχουμε το δεύτερο τμήμα. Της 196. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 197 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Συμβιβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 234 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.38 Donjon, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.39 δεν ψηφίζουμε γλωσσική τροπολογία. 2.40 φώτιγκα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φώτικα 267 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2,69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2,70 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε φύτο, τροπολογία 2,70. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται, ευχαριστώ. 2,71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Να το ελέγξουμε. Μποστινάρου τροπολογία 279 ψηφίζουμε τώρα. Να σηκώνετε καλύτερα τα χέρια σας παρακαλώ. 2.80. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27. Υπέρ κατά... Να θέλετε να το ελέγξουμε. Να ψηφίσουμε τη 2.80. Εντάξει, ψηφίζουμε τη 2.80 ηλεκτρονικά. Τη 2.80. Πέντε μέλη δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Καλώς πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όπως το είπα. Συμβιβαστική 27. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.95. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έτσι δεν είναι. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 305. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 306 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3,58 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε, να ψηφίσουμε την 308. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κάποιοι από εσά δεν ψηφίζετε. 309 κατά πίπτη 310 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ψηφίζουμε την 310 παρακαλώ η 309 κατά πίπτη την 310 ψηφίζουμε I close the vote. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 3.11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 3.13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.16. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 325. Από την 3.15 μέχρι την 3.32 λέει η Πρόεδρος. Όχι. Δεν συμφωνείτε. Άρα μία-μία θα τις ψηφίζουμε. Πάμε και να ψηφίσουμε την 3.25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 328 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 329 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε την 330 καλώς ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 330 παρακαλώ Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 3.31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3.33 της κυρίας Φώτιγκα. Υπέρ, κα, κατά, αποχές εγκρίνεται 3.34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3.35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3.36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3.37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 3.38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις recital υπαριθμών 7. Κέλαμ, όλες είναι από την 7 μέχρι την 11, να τις ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συγχαρητήρια κύριε Κέλαμ. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην αιτιολογική σκέψη α μεγάλο και α μικρό 23, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 25 ηλεκτρονικά. Άλλη φορά να σηκώνετε καλύτερα και περισσότερο τα χέρια σας. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 25, παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 κυρία Φώτιγκα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 Μποστινάρο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 56 καταπίπτει, 57. Όχι, δεν καταπίπτει. Ναι, καταπίπτει αν εγκρίθηκε η 54. Όχι. Ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε την 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα θα, την, θα το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 56. Παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορείτε να σηκώνετε τα χέρια σας καλύτερα. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. 63 μάλλον. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58, ελέγχουμε. 68, όχι συγγνώμη, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 67. Την 67 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές Γκόμες. Ψηφίζουμε τροπολογία Γκόμες 76. Παρακαλώ. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 87, όχι, συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 87 αποσύρθηκε, 102 ΠΑΕΤ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 103 Φώτικα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 104 καστάλτο. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, citations, αιτιολογικές αναφορές, προφορική τροπολογία υπαριθμών 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αριθμός 1, σάκε, πάετ κλπ.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 Τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε ψηφίσμου ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία για το σύνολο της έκθεσης τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Κούζο, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από πλευρά Γκουε θα υποβάλουμε έκθεση μειοψηφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούζο.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 Είχαμε μια αλλαγή στο πάνελ. Να περάσουμε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ο κύριος Πάσκου είναι ο εισηγητής. Και τώρα να ψηφίσουμε. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, να κρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 117 και 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 120. Έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εάν δεν σηκώνετε τα χέρια σα, θα χρειάζεται να κάνουμε διαρκώ ελέγχου. 121. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 133. Μαρί. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 147 αντάκτουσον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι θέλετε να κάνω έλεγχο 147 147 έλεγχος ηλεκτρονικά πέρας της προφορίας απορρίπτεται Σοφοζέρ 148-149 Ταυτόσιμε. υπέρ, κατά, εποχέ, απορρίπτονται 150 υπέρ, κατά, εποχέ. απορρίπτονται Απορρίπτονται. 151 υπέρ, κατά, εποχέ. Απορρίπτονται. 152 υπέρ, κατά, εποχές απορρίπτονται. 153 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 154. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155. Υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. 156. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157. Έλεγχος για την 156. Να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε. 162. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 απο, αποσύρεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 198 Καστάλντο. Πέρας. Βλέπετε, Απορρίφθηκε τελικά. Δυστυχώ, κύριε Καστάλντο. 199 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε και αυτήν. 199. Θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο αν δυσκόνται τα χέρια σας. Νομίζω εγκρίνεται. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.16, 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ έλεγχο και 217, 217 έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Γιατί δεν ψηφίζετε, μας λείπουν δύο. Τρίφ. Πέρας. Εγκρίνεται. 100, μάλλον 218 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 219 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 231-232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Για να ελέγξουμε 231-232. Δεν είναι σαφές. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω. Μας λείπουν δύο. Πέρας. Βλέπετε, απορρίφτεται. Διότι δύο από εσά δεν είχαν ψηφίσει. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 243 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 246 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 247 υπέρ κατά ξανά. 247 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για τη 247. Δεν είναι σαφές. Πέρας. Απορρίφθηκε. Σοφοζέρ 248 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 249 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 250 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 250, ναι. Θέλετε έλεγχο. Ωραία. Έλεγχος για 250. Πέρας. Εγκρίνεται 251 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 252 απορρίφ, αποσύρθηκε, οπότε δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Δεν ψηφίζουμε την Μανέσκου 252. 253 253 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Συμβαστική 17, 15. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 261-262 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 270 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ε, απορρίπτεται. 271-273 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, 272 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 274 υπέρ κατά αποχές 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 275 υπέρ κατά αποχές 275 Καστάλντο. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 275. Πέρας. Απορρίπτεται. 276 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 277 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 278 αποσύρεται, αποσύρεται. 280. Ε, 280 υπέρ. Συγγνώμη. Τι μου λέτε. Τη 277. Ωραία. Ε, εντάξει, ας την ελέγξουμε. 277. Πέρας. Ευχαριστώ. 280 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 281 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σοφοζέρ 298. 298 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 299 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 300 αποσύρεται. 301 υπέρ, 301 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα 302, 303, 304, 305 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 306. 311. 311. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. Και τώρα 338, σοφοζέρ και πάλι, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 339 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 342 υπέρ κατά αποχές έλεγχος απορρίφθηκε μάλλον. 343 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 344 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητηρία. Συμβεστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 347-348 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 349-350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 351 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 352 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 356 υπέρ κατά αποχές να κάνουμε έλεγχο. Πρέντα, 356. Μας λείπουν τρεις. Ε, okay, I close the vote. Πέρας. Εγκρίνεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 359 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, λογική σκέψη ε, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα και πάλι στη, στον κύριο Σοφοζέρ 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές 55 υπέρ, κατά, αποχές, βίστησε να ελέγξουμε για την Αντιπρόεδρος. Να είμαστε βέβαιοι. Τρεις μας λείπουν. Δύο λείπουν τώρα απορρίπτεται, αλλά με μικρή διαφορά.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 Κανείς δεν συμμετέχει. Κοιμάστε. Μας λείπουν πέντε. Πέντε ψήφοι. Δεν θέλετε να ψηφίσετε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83. Α, 84. 84 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, Κύριε Φρόιν, πρέπει να κάνω έλεγχο. Κανείς δεν σηκώνει τα χέρια του. Πέντε ψήφοι μας λείπουν. Επίτηδες το κάνουν. Πέρασε τη ψηφοφορία σου. Εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω. 94 έλεγχος για την 93 ωραία λοιπόν έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος Μποστινάρου 97. Δεν είναι σαφές. Πέρας. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Να κάνουμε έλεγχο για την 98. 98 έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές 1 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 4 4 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 6. Έλεγχος παρακαλώ. Κάτι περιμένετε φαίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, καταπίπτουν. Καταπίπτουν και οι 7 και οι 8. Και τώρα, τελική ψηφοφορία για την έκθεση όπως τροποποιήθηκε. Μας λείπουν διάφοροι. Μας λείπουν πέντε ψήφοι, σας παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Πάσκου. Ωραία. Προχωρούμε. Τώρα πάμε στο 10. Σημείο 10. Έκθεση Γκέρενς. Σημείο 10 παρακαλώ. Να συνεχίσουμε αμέσω. Προ μια εξωτερική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των προήμων και καταναγκαστικών γάμων, επόμενα βήματα.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 167 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 165, όχι, καταπίπτει. Συγγνώμη, συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 Μόμπαρικ. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ δύσκολε οι ψηφοφορίε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ψηφίζετε τις δεν μετράτε τις ψήφους, ε, απλά κοιτάτε με το μάτι πόσα ε, χέρια σηκώνονται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σέβεστε περισσότερο τη διαδικασία, διότι με βάση ε, τον κατάλογο των ψηφοφοριών κρίνεται αυτό είναι δημοκρατία. Ο κόσμος πληρώνει για όλα αυτά. Μας ζητάτε να σηκώσουμε το χέρι μας, αλλά ε, διαβάζεται πολύ γρήγορα, λίγα δευτερόλεπτα μόλις ε, κρατάει όλη η διαδικασία, κανείς δεν έχει καταλάβει που βρισκόμαστε. Περί παροδίας πρόκειται. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ξέρετε ότι έχουμε συμβαστικέ προτάσει. Όλη η δουλειά έχει γίνει σε συναντήσει των σχεδόν εισηγητών ε, και τι επιτροπέ. Όχι, τσίρκο είναι εδώ. Κάθε ψήφος μετράει. Δημοκρατία έχουμε. Αλλιώς θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά κάθε φορά. Ε, πρόεδρος, ε, ναι, μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε. 196. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΦΑΜ 13. 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 220 είκοσι. Μπούχνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το επαληθεύσουμε. 227. Uh, we miss some Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Τρεις ψήφοι λοιπόν. Ωραία, ας προχωρήσουμε. πέρα τη ψηφοφορία. απορρίπτεται. 226 υπέρ. Κατά αποχές, Απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. 229 ηλεκτρονική επαλήθευση. Για να είμαστε βέβαιοι. It's... I close the vote. Πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Σα ευχαριστώ που σήκωσα τα χέρια σα. 231 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. ΦΑΜ 19 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 24 της Επιτροπής Γυναικών, όχι αυτή είναι απαράδεκτη. Ε, έχουμε το θέμα του απαράδεκτου. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Μπορώ να προχωρήσω, ωραία. Αιτιολογική σκέψη α, ε, συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35, 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26. Ηλεκτρονική επαλήθευση. I close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. Μία ψήφος έλειπε. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, τότε γιατί δεν τα χέρια. ψηφοφορία. close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Okay, we know now. Compromise. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Αιτιολογική σκέψη G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίν, ε, αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Φαμ ο, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ τ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φαμ Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 3 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 6. Ελέγχουμε την 6. Adopted. I close the vote. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί. Δύο ακόμα πρέπει να ψηφίσουν. πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε στο σημείο 11. Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γεών. Προχωράμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. We have a lot to do. Παρακαλώ συγκεντρωθείτε, έχουμε πολλή δουλειά. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 δεν ψηφίζουμε. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 αντάκτουσον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 επαλήθευση Ζέλερ κλπ.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 λέει η πρόεδρος. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. 137. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 139. Καταπίπτει. Και 138. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 144. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 145. Υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 145. Απορρίπτεται νομίζω. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε. 146 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 147 δεν ψηφίζουμε. 148 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ποιο... Ποια θέλετε να ελέγξουμε. Συμβαστική 15 ψηφίσαμε. Συμβαστική 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα 168 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 168 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε παληθεύσουμε την 171. Άλλοι 7 πρέπει να ψηφίσουν. Έξι ψήφοι. Δεν θέλετε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 172. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται ε, κοιτώντας τα χέρια, αλλά ηλεκτρονική επαλήθευση. 173. Six votes are missing. Έξι ψήφοι λείπουν. Okay, now we close the vote. <laughs> Thank you. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 να το ελέγξουμε. Θέλετε να ψηφίσουμε τη 203. Ψηφίζουμε λοιπόν τη 203. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 205. Την ψηφίσουμε λοιπόν. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ. Καλώς. Λείπουν τρεις ψήφοι, αλλά εν περιπτώσει εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.11 υπέρ κατά απορρίπτεται να το ελέγξουμε θέλετε να το ελέγξετε εντάξει καλώς ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 2.11 Πέντε δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αλλά με το μάτι δεν φαίνεται, δεν είναι καθόλου σαφές. Θέλω να τα κάνω σωστά. σωστά. 2-12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιατί να το ελέγξουμε ε, τη 2.12 κύριε Μπούχνερ αφού την εγκρίναμε την τροπολογία σας. Θέλετε να το ελεξουμε Καλώς, 2.12 ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δύο, ένα, τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ψηφίσουμε πάλι. Καλώς. Πέντε ψήφοι λείπουν. Δύο δεκατέσσερα ψηφίζουμε. Τη δύο δεκατρία εγκρίναμε. Υπέρ δύο δεκατέσσερα κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε τη 2.14. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω χρόνο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 2.14. Καλώς. Πέντε ψήφοι λείπουν πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Να ξέρετε ότι είναι πέντε που δεν ψηφίζουν. Συμβιβαστική 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.21. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές θέλετε να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Καλώς. Την 11 ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη που ψηφίζουμε τόσο πολύ ηλεκτρονικά. 5 δεν ψήφισαν. Πέρα στις ψηφοφορίες. Τρομερό. Συμβιβαστική 27. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα του 17. Καλώς. I close the vote. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Free vote. 42. Υπέρ. Τη 41. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 41. Καλώ ψηφίζουμε τη 41. Πέρας. Απορρίπτεται. 42. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές 43 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τη 43. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές θέλετε να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 45. Ψηφίζουμε τη 45. We close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 δεν ψηφίζουμε. 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές δεν, δεν είμαι βεβαία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 61. 62 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. 53. Θέλετε να ψηφίσουμε την 54. Καλώς. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Και τώρα η 53 καταπίπτει. Συμβιβαστική 36. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 71 τώρα. Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη. Πάμε στην 71. Καλώ, συγγνώμη. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 73. Ελέγχουμε την 73 παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Όχι, 75. Καταπίπτει. 76. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, 79. 79 απορρίπτεται. Νομίζετε, δεν είμαι βεβαία, θα, δεν θέλω λάθη, θα το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεν θέλω να παραπλανήσω κανέναν. Ψηφίζουμε την 79 παρακαλώ. «48 είναι παρόντες και πάντοτε έχουμε 45 ψήφους. Δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει. Εγκρίνεται. Δεν με αφορά εμένα. Υπαριθμόν 1, citation 3. Υπέρ κατά αποχές 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά υπαριθμόν 2. Την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Citation 2. Πέρασε. απορρίπτεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, 5. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για την 5 λοιπόν. Θέλετε να, ψη... να ελέγξουμε την 5. Καλώς. Ψηφίζουμε την 5. We close the vote. Adopted. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ερχόμαστε στη τροπολογία από την Επιτροπή ΦΕΜ 1. Καταπίπτει. Τη 2 της ΦΕΜ, της Επιτροπής Γυναικών. Υπέρ. Κατά αποχές της ΦΑΜ 2. Γυναίκες 2 από την Επιτροπή αυτή. 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ 3 πρώτο τμήμα κατά τμήματα. Καταπίπτει το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τρίτης τροπολογίας από την Επιτροπή για τις Γυναίκες. Μόνο το δεύτερο τμήμα του ΦΕΜ 3 δηλαδή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Γιατί να το ελέγξουμε. Εντάξει, θέλετε να το ελέγξουμε. Το ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3 από τις ΦΑΜ. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 4 της ΦΑΜ. Πρώτο τμήμα. Καταπίπτει. Δεύτερο τμήμα μένει. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος της τροπολογίας 4 από την Επιτροπή για τις Γυναίκες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν με πιστεύετε. Καλώς, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της ΦΑΜ 4. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5. Από τη γνωμοδότηση της ΦΑΜ. Καταπίπτει και το 6 και το 7. Πάμε στο 8. Ψηφίζουμε το 8 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 9. Τώρα με πιστεύετε. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Ποιος θέλει να το επαληθεύσουμε. Το 9. 9 από φαμ. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σίγμα υπέρ, τι θέλει να ελέγξουν. Ποιο θέλει να έλεγξουν. Το ε, την εταιρεολογική σκέψη ε, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αποφάμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπουν έξι ψήφοι. Αν κοιμούνται δεν μας ενδιαφέρει. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η αιτιολογική σκέψη ε. Σίγμα ταφ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ζ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λάμδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μη υπέρ τίποτα. Η όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το Q τελευταία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη γνωμοδότηση DEVE, υπαριθμών 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 1 της DEVE, κύριε Πρέντα. Ό,τι πείτε. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Είχατε δίκιο κύριε Πρέντα και σας ευχαριστώ. ΔΕΒΕΤΡΙΑ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το ελέγχουμε. Το επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 4. Δεν είναι η ίδια πλειοψηφία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 5. Κα, υπέρ, κατά. ΔΕΒΕ 5. Υπέρ, κατά. Αποχές. Το επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 5 ΔΕΒΕ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεβε 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεβε 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεβε 8. Πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Καλώς. Δεύτερο τμήμα της ΔΕΒΕ 8 ψηφίζουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην ΔΕΒΕ 10 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας, συγγνώμη. Πρώτο τμήμα της ΔΕΒΕ 10. Πίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. καταπίτη ΔΕΒΕ 11. Υπέρ. Κατά αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ΤΕΒΕ 11. Δεν είναι η ίδια πλειοψηφία. Δεν είναι. Το παρακολουθούμε στενά και δεν είναι η ίδια. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 τίποτα. ΔΕΒΕ 13. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλώς, το ελέγχουμε. Εσάς κοιτάζω κύριε Ράιλι. Τι πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 15, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. ΔΕΒΕ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Την 25, ΔΕΒΕ. Παρακαλώ, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται δεν είναι η ίδια πλειοψηφία. ΔΕΒΕ 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει. ΔΕΒΕ 31. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και εξηγήσει μετά την ψηφοφορία θα υπάρξουν. Ρωτάει ο βουλευτή. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την υπομονή σα και τη συνεργασία σα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο το εγχείρημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Now there is no break. Give maybe one minute. Only one minute break for those who want to leave. Κανένα διάλειμμα, ένα λεπτό μόνο για όποιον θέλει να βγει και να συνεχίσουμε με το σημείο 12, την κατάσταση στην Αρμενία. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll have to continue. Now we proceed to the exchange of views on the situation in Armenia. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τώρα με την ε, κατάσταση στην Αρμενία. Ξέρετε ότι ακολουθήσαμε τη διαδικασία της συνένεσης για την ε, συνολική και ενισχυμένη συμφωνία συνεργασίας με την Αρμενία, για την οποία ψηφίσαμε νωρίτερα σήμερα ίσχυση. Έχει ήδη αυτό ολοκληρωθεί στην Επιτροπή μας και ξέρετε ότι την προερασμένη εβδομάδα στις 8 Μαΐου ο κύριος Πασινιάν εξελέγει από την Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας Πρωθυπουργός. Αυτό μετά από δύο εβδομάδες διαμαρτυριών στο Γερεβάν κυρίως και οι διαμαρτυρίε αυτές ήταν ειρηνικέ με τη συμμετοχή βουλευτών και ακτιβιστών για την, μετά την παρέτεση της 24 Απριλίου ε, του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου κυρίου Σαρκισιάν. Στις 24 Απριλίου οι πρόεδροι αυτής της Επιτροπής και της Διακοινοβουλευτικής ε, Συνέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξέδωσαν μία ανακοίνωση μετά την εκλογή της 8 η Μαΐου. Ο πρόεδρος Μακάλιστερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Πασίνιαν ε, στην σημερινή συνεδρίαση. Δυστυχώς δεν μπορούσε να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες για λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Οπότε μπορούμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Τατούλη Μαρκάριαν, ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην Αρμενία που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση των πραγμάτων εκεί. Να δώσω το λόγο στην εξοχότητά του στον κύριο Μαρκού Μαρκέριαν, ε, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο. Α, θα μείνετε εκεί που είστε. Εντάξει, θα πάρτε το λόγο από εκεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, επειδή σήμερα μιλάμε για τη δημοκρατία της Αρμενίας και τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εκεί πρόσφατα, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώντας προηγουμένως τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που έδωσαν τη συνένεσή τους στην ε, ε, έγκριση τη συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ε, Δημοκρατία τη Αρμενία. Όπω ξέρετε, η Δημοκρατία τη Αρμενία ομόφωνα έχει εγκρίνει την συμφωνία και την προσωρινή τη εφαρμογή, η οποία θα ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου 2018. Ε, όπως έχει ήδη δηλωθεί επανειλημμένως, η ιουνιου 2018 οπω αποδίδει μεγάλη σημασία στην εμπάθηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτήν την έννοια, η σύντομη έγκριση και κύρωση της ε, συνολικής και ενισχυμένης συμφωνίας εταιρικής σχέσης με τη Δημοκρατία της Αρμενίας και ε, με μεταξύ αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα έγγραφο που δείχνει τη δεσμευσή μας στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα με μια σταθερή βάση για να ενισχύσουμε τον πολιτικό μας διάλογο στο πλαίσιο της οικονομικής ε, συνεργασίας και της συνεργασίας ασφαλείας καθώς και την κινητικότητα των πολιτών μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με το καθεστώς απελευθέρωσης θεωρήσεων και το σχετικό διάλογο. Ελπίζουμε ότι η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι ένα θετικό μήνυμα και προ τα κάτι μελη για να επιταχύνουν την διαδικασία κύρωση. Η νέα αυτή συμφωνία μαζί με τι προτεραιότητε εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία νομίζω ότι θα δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνεργασία μα και θα φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για του πολίτε μα. Κυρίε και κύριοι, Όντω, η νέα Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία για τι διμερεί μα σχέσει είναι ένα σημαντικό θέμα και σοβαρό θέμα για συζήτηση. Υπ' αυτήν την έννοια, το να συζητήσουμε τι πρόσφατε πολιτικέ εξελίξει στην Αρμενία είναι ε, εύστοχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργό ρόλο στην ε, θεμελίωση τη δημοκρατία στην Αρμενία. Οι πρόσφατε εγχώριε πολιτικέ εξελίξει έδειξαν ότι ο κόσμος της Αρμενίας ε, παίρνει την, ε, τα ιδεώδη της δημοκρατίας πολύ σοβαρά και είναι αφοσιωμένο ε, στην προάσπιση του. Δεν θα μπω στι λεπτομέρειε των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων, αλλά σήμερα, καθώ η πολιτική κρίση βρίσκεται πίσω μα, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι καθ' όλη αυτή την περίοδο οι πολίτε τη Αρμενία ελεύθερα εξάρχισαν τα δικαιώματά του με ειρηνικό και μη βίαιο τρόπο. Όλες οι πλευρές έδειξαν αυτοσυγκράτηση με έναν ουσιαστικό διάλογο να δημιουργείται ώστε να μπορέσει ειρηνικά να διαδηλώσει ο κόσμος του δρόμου του Γερεβάν και βάσει του συντάγματος της Αρμενίας να περάσει εξουσία σε άλλα χέρια. Αυτό δείχνει το υψηλό επίπεδο πολιτικής οριμότητας που έχει πετύχει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η δημοκρατία και η πορεία εκδημοκρατισμού της Αρμενίας είναι πλέον ε, αμετάκλητη. Η νέα κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί προς το στόχο αυτό και να έρθει ε, σε ευθυγράμμιση με τις ε, βέλτιστε πρακτικέ τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κυβέρνηση του κυρίου Πασινιάν ε, συμμετέχουν επαγγελματίε ε, και εμπειρογνώμονε από όλα τα πολιτικά κόμματα. Κυρίε και κύριοι, αναμένουμε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα σε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια για να εκπληρώσουμε τι προσδοκίε και τι μεγάλε ανάγκε των κοινωνιών μα. Εγώ θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να εκφράσω την την ευχαριστία μας τις ευχαριστίες μας προς την διαρκή, ε, για τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του Ευρωκοινοβουλίου, ε, της Επιτροπής αυτής εξωτερικών υποθέσεων, της διακοινωνιστικής συνέλευσης, ε, που προσφέρουν όλη τους τη στήριξη στη Δημοκρατία της Αρμενίας, ώστε να μπει στη σωστή πορεία εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για αυτήν την ε, ενημέρωση. Βλέπω εδώ τον κύριο Τόκες που είναι μπροστά σας. Επειδή είναι εισηγητής ε, για τα θέματα της Αρμενίας, νομίζω ότι θα μπορούσε να προσθέσει κάτι. Έχετε το λόγο. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Πρόεδρε, σήμερα η Επιτροπή αυτή ψήφισε συντριπτικά υπέρ να συνενέσει το Ευρωκοινοβούλιο στη νέα συνολική και ενισχυμένη συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκής... της ε, Δημοκρατία τη Αρμενία. Αυτό ήταν μεγάλη χαρά για μένα που υπήρξα συγητή ε, για τα θέματα τη Αρμενία. Επειδή ανέλαβα την εκπόνηση τη ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου με σκοπό τη συνένεση και το συνοδευτικό ψήφισμα. Ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους μου για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε καθ' όλη την ε, διαδικασία αυτή στην Επιτροπή, καθώς και τη Γραμματεία για τη στήριξή της. Και τους συνεργάτες της ομάδας μου, την Τζουλιάνα και τον Ρόμπερτ. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την Αρμενία, τα, οι τα δραματικά γεγονότα που εξελίχθηκαν παράλληλα με την εξέταση της ε, συμφωνίας από την Επιτροπή μας απασχόλησαν πολύ το Κοινοβούλιο και ακόμη απασχολούν και σήμερα. Στην έκθεσή μας επικροτήσαμε τους πολίτες της Αρμενίας και την ε, αλλαγή ε, εξουσίας με ειρηνικό τρόπο σε επίπεδο κυβέρνησης και βάσει του συντάγματος και επίσης καλωσορίσαμε την αυτοσυγκράτηση που έδειξαν οι δυνάμεις δίωξης ε, ε, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Αλλά όπως είπε σύντομα και η Πρόεδρος, επίσης μας απασχολεί ο αριθμός συλλήψεων ειρηνικών διαδηλωτών συμπεριλαμβανομένων ε, ε, Αρμένιων βουλευτών. Καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε ότι σήμερα ακόμη 41 άνθρωποι ε, αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ποινικέ κατηγορίες και ίσως είναι η στιγμή να αναθεωρήσουμε το άρθρο 225 του ποινικού κώδικα για την διοργάνωση μαζικών διαμαρτυριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρχές, αλλά θα ήθελα να ζητήσω και από τον πρέσβη Μαρκαριάν να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις υποθέσεις και επίσης να μεταφέρει τις ανησυχίες μας στους υπευθύνους του Γερεβάν. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας <clears throat> ότι οφείλουμε συγχαρητήρια στον κύριο Πασινιάν για την εκλογή του ως Πρωθυπουργού της ε, Αρμενίας και παροτρύνουμε την κυβέρνησή του με βήμα ταχύ να προχωρήσει στην εκπλήρωση των προσδοκιών των Αρμένιων πολιτών. Όλος ιδιαίτερος ως προς το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως αναφέρει και η έκθεσή μας, η Επιτροπή αυτή και βεβαίως ολόκληρο το Ευρωκοινοβούλιο αναμένουν διακαώς την ενισχυμένη συνεργασία με την Αρμενία, τους πολιτικούς της ηθήνοντες και την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τόκες για τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, στον κατάλογο μου έχω πέντε συναδέλφους που θέλουν να, να τοποθετηθούν. Εάν θέλει κι άλλος κανείς το λόγο, θα κλείσουμε τώρα τον κατάλογο των αγορητών, να μου το πείτε. Σε αυτούς τους πέντε θα δώσω το λόγο για ένα δίλεπτο στον καθένα. Η κυρία Μούντι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη που ήρθε εδώ σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπε ο προλαλής σας, ότι ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα σήμερα το πρωί. Υπάρχει όμως και η συμφωνία ΣΥΠΕΡ και θα ήθελα να σχολιάσω επίσης το, το δημοκρατικό πνεύμα που ήταν προφανές πρόσφατα στην Αρμενία. Και οι συνέπειες του φάνηκαν στην εκλογή του κυρίου Πασινιάν. Πού βρισκόμαστε τώρα, τι έχει προταθεί σχετικά με μελλοντικές εκλογές. Θα ήθελα λοιπόν μια ενημέρωση από εσά σχετικά με τα επόμενα κοινοβουλευτικά βήματα, κατά τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Τόκεσε και να εκφράσω την υποστήριξη της Επιτροπής μας στην Συνολική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρέσβη για αυτά που μας είπε για την Αρμενία. Για λόγους που πολύ καλά καταλαβαίνουμε, η Αρμενία θα πρέπει να είναι χώρα στην οποία θα πρέπει να αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους τους τομείς που δεν εμπίπτουν στην DCFTA, στην ε, συμφωνία αυτή, θα πρέπει να βρούμε ρύθμιση. Ε, σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε και θετικό αποτέλεσμα στην Ολομέλεια. Η Αρμενία ε, έχει δείξει ότι είναι όριμη δημοκρατία, ε, σέβεται την δύναμη του λαού αλλά εντός του κράτους δικαίου. θα επικροτούσα περισσότερες ευκαιρίες ε, προς τους ε, Αρμένιους πολίτες να επισκεφτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκεφτούν την Αρμενία που είναι αρχαίος και πλούσιος πολιτισμός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέτινα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας, διότι θα μιλήσω τσέχικα. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τόκες που κατάφερε να ενημερώσει ε, να επικαιροποιήσει την έκθεσή του και να συμπεριλάβει ακόμη και τα πιο πρόσφατα γεγονότα τα οποία είδαμε στη Γερεβάν και άλλες πόλεις της Αρμενίας. Ε, είδαμε πόσο σοφός είναι ο λαός της Αρμενίας. Ε, δεν... Ε, υπέκυψαν και είδαμε μια δημοκρατική μεταφορά της εξουσίας στην Αρμενία. Η Αρμενία λοιπόν έχει αποδείξει ότι είναι έτοιμη να χειριστεί τη σύγκρουση ανάμεσα στην ε, Αρμενία και το ε, Αζερβαϊτζάν και να δώσει τέλος σε αυτήν. Ε, ελπίζω ότι έχει ανοίξει πια ο δρόμος, ώστε ε, να βρεθεί η λύση. Το αξίζει η ανεξαρτησία στο Ναγκόρνο Καραμπάκ και θα πρέπει να αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από άλλους ηθινόντες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέτινα. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Πρέσβη που ήρθε εδώ σήμερα να μας ενημερώσει. Με πολύ αγωνία παρακολουθήσαμε την ε, ειρηνική αυτή μεταφορά της ε, εξουσίας ε, στην Αρμενία, στο στη Γερεβάν. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση, διότι το νέο Αρμενικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε ομόφωνα την νέα συμφωνία μόλις πριν ξεδηληθούν τα γεγονότα αυτά και Πιστεύω ότι ε, έχουμε έναν πολύ καλό οδικό χάρτη με την ε, Συμφωνία ΣΕΠΑ και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αυξήσει την ε, ενίσχυσή της προς τον προϋπολογισμό, προς την δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις αυτές υπό την καθοδήγηση της νέας κυβέρνησης. Θέλουμε όμως μια επικοδομητική προσέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει στην ε, Αρμενία ε, πολύ ισχυρή πόλωση, όπως είδαμε στη Γεωργία, κάτι που δεν έχει βοηθήσει τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Γεωργίας. Μιλώ ως επικεφαλής της αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την ε, παρατήρηση των ε, εκλογών πέρσι και η νέα κυβέρνηση θέλει να οργανώσει πρόορες εκλογές και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε εγκαίρως την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, παρατήρηση των εκλογών, διότι είδαμε τι έγινε την προηγούμενη φορά, είδαμε εκφοβισμό των ψηφοφόρων ε, και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόρτη, λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ ήμουν στην αποστολή για τις εκλογές ως παρατηρητή στην Αρμενία και πρέπει να σας πω ότι η πολιτική αλλαγή είναι σημαντική. Δεν μπορούμε όμως να θεωρούμε ότι η υπερδιαρθρωτική αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας είναι και η λύση στα προβλήματα της Αρμενίας. Οι εκλογές που έλαβαν χώρα ε, ήταν εξαιρετικά ανησυχητικές, όχι μόνο για το τυπικό θέμα της για ό,τι φαίνεται, αλλά για το λανθάνον θέμα, αυτό που υπάρχει στην κοινωνία της Αρμενίας, που υπάρχει από την παθολογία μιας χώρας που έχει ένα πληθυσμό που συνεχώς μειώνεται και δεν αυξάνεται γιατί η νεολαία μεταναστεύει. Η νεολαία δεν έχει μέλλον στη δική της χώρα, στην Αρμενία και συνεχώς μεταναστεύει. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Αρμενία έχει χωριστεί σε ολιγαρχικές ομάδες που ελέγχουν ε, την οικονομία με τρόπο κατακαιρματισμένο. Δεν είναι θέμα μόνο η διαφθορά που είναι τεράστιο πρόβλημα. Εγώ εύχομαι το καλύτερο για τον αρμενικό λαό και ελπίζω να μπορέσουν να προχωρήσουν και να λύσουν τα προβλήματά τους, αλλά να μην περιοριστούμε απλά να εκφράζουμε ικανοποίηση γιατί άλλαξε η κυβέρνηση, ενώ δεν έχουν αλλάξει οι συνιστώσεις οι κοινωνικο-οικονομικές και οι κοινωνικο-οικονομικές σταθερές που είναι οι, οι, θεμελιώδεις. Αλλάζουμε την επιφάνεια και δεν αλλάζουμε τη δομή, τα θεμέλια που βασίζονται στην ολιγαρχία και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα και όσο περιμένουμε αυτά τα ολιγαρχικά θεμέλια η Αρμενία δεν πρόκειται να προχωρήσει και να προοδεύσει. Καλό θα ήταν να είχε μεγαλύτερη οικονομική εγκύτητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω όμως τα στρατηγικά της προβλήματα και μάλιστα την ανάγκη παρουσίας ε, ε, ασφαλείας από την Ρωσία. Δεν το λέω για να το απορρίψω, ούτε να απορρίψω τη δική μας θέση. Πρέπει κανείς να καταλάβει ποια σχέση έχει η Αρμενία. Νιώθει σαν σάντουιτς, νιώθει πιεσμένη ανάμεσα στην Τουρκία και στο Αζερβαϊτζάν. Όμως δεν μπορεί να είναι και επιμονή μου βάση ως ε, φυλακισμένη σε αυτή τη σύγκρουση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Δεν τους βοηθά αυτό να λύσουν τα προβλήματα τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Καρστάλτο παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω ξανά τον ε, πρέσβη για την παρουσία του εδώ και τις πληροφορίες που μας έδωσε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Τόκιος για τη δουλειά του. Αυτό που συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες είναι ξεκάθαρα μια ιστορική ε, εξέλιξη σημαντική για την ε, δημοκρατία της Αρμενίας. Όμως πρέπει να το θεωρήσουμε απλώς ένα πρώτο βήμα. Ένα πρώτο βήμα για τις περαιτέρω προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Πιο συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προταθεί από τον νέο Πρωθυπουργό, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, η διοργάνωση νέων βουλευτικών εκλογών σύντομα, όπως ζήτησε ο Πρωθυπουργό, και άλλες προκλήσεις που έμειναν αναπάντητες εδώ και πολλά χρόνια, όπως ε, κάποια αποφασιστικά βήματα κατά της διαφθοράς και η αποσάρτρωση, ε, των, η διάλυση αυτών των ελίτ, των ολιγαρχιών που έχουν ε, δυσκολέψει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, όπως και σε άλλες γειτονικές είναι σημαντικό αυτό για την γειτονία μας, για την γειτονία μας ιδίω στην Νότια και για αυτόν τον λόγο πρέπει κάπως να αποδομήσουμε αυτού του είδου τα δίκτυα και τα συστήματα για να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει μια οικονομική αναγέννηση και να πάυσει αυτή η διαρκής διαρροή εγκεφάλων και ταλέντων προς το εξωτερικό. Είναι σημαντικά για να ε, χτιστεί το μέλλον τη χώρα. Και θέλω ξανά να τονίσω και να θυμίσω την ανάγκη να είμαστε από πλευράς μας διαρκώς ε, δίπλα στον ε, λαό της Αρμενίας, την πορεία του αυτού και πρέπει να ξαναρχίσει και η προσπάθεια ερήνευσης με το Αζερβαϊτζάν, να ξεφύγουμε από τα πλέγματα των τελευταίων ετών και να ε, πούμε και στην ύπατη εκπρόσωπο ότι το πλουστάσιο η φαρέτρα εργαλείων που έχουμε στη θέσή μας για να προωθήσουμε τις σχέσεις μας με την Αρμενία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είμαστε λοιπόν σύμμαχοι και φίλοι στη διαδικασία αυτή και ελπίζουμε σύντομα να δούμε περαιτέρω μηνύματα ενθάρρυνσης, ιδίω στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Αστρεβίτσιος. Και μετά έχει κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον πρέσβη για τη σημερινή ενημέρωση. Ήθελα να τονίσω από την πλευρά της συνεργασίας Ευρωκοινοβουλίου με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας ότι η στιγμή αυτή αλλαγής, πολιτικής αλλαγής στην Αρμενία ήταν μια θετική εμπειρία και επίσης και ένα δείγμα, ένα μήνυμα για την ευρύτερη γεωγραφική ζώνη καθώς δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες δημοκρατικών ε, μεταβάσεων στις χώρες της γειτονίας μας. Άκουσα μάλιστα ε, συγκεκριμένες πληροφορίες από το Γερεβάν και άλλα μέρη στην Αρμενία και το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολίτες οι ίδιοι ανέλαβαν την ευθύνη της αλλαγής. Η Σιτουαγιά ε, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό την κατάλληλη στιγμή, ακριβώς όταν έπρεπε, αποφάσισε να παρατηθεί. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει αλλαγή και στην Αρμενία, αλλά σε αυτήν την χρονική στιγμή ήταν κάτι πολύ θετικό αυτό για τη δύση της Υπήρου μας. Και τώρα η κατάσταση βεβαίω στο Κοινοβούλιο, στη Βουλή σα είναι κάπω προβληματική, υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία των τελευταίων εβδομάδων και το δίδαγμα ε, για τα σφάλματα, τα διδάγματα από τα σφάλματα του παρελθόντο, θα σας δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε την πολύ δύσκολη κατάσταση του Κοινοβουλίου. Δεν είναι εύκολο αν μια κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αλλά ελπίζω ότι θα δούμε επικοδομητική εξέβρεση λύσεων όπως είδαμε να συμβαίνει τις προηγούμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και πραγματικά ξαναλέω ότι είναι η τελειότερη στιγμή αυτή. Η στιγμή που επέλεξε ο κύριος Αρκισιάν για να παρατηθεί. Καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό για την Ευρώπη και καλό για την Αρμενία. Ο κύριο Αστρεβίτσιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλωσορίζω τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αρμενία. Είναι ο σωστός τρόπος, η σωστή κατεύθυνση. Και ε, επειδή είχαμε ειρηνικές διαδηλώσεις στην Αρμενία, στους δρόμους, όπου επικεφαλής ήταν ο κόσμος οι άνθρωποι, οι πολίτες. Είναι αυτοί που ξέρουν ποιε αλλαγέ χρειάζεται μια χώρα και αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για του πολιτικού που προσπαθούν να χειραγωγήσουν του πολίτε και να επιβάλλουν συνταγματικέ αλλαγέ. Από το 2015 οργανώνουν δημοψηφίσματα, ενώ ήδη από τότε ακούγονταν φωνέ δημορτυρία. Αυτό μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για παραπλάνηση και προσπάθεια να χειρολογηθούν οι πολίτε με πληροφορίες που δεν γνώριζαν. Η Αρμενία λοιπόν έχει κάνει ένα σωστό βήμα. Χρειάζεται και άλλη οικονομική και κοινωνική ε, πρόοδο βεβαίω, να έρθει σε ένα νέο επίπεδο η οικονομία και η κοινωνική προστασία. Και χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει σε αυτή τη συνολική Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Είδατε ότι εγκρίθηκε με πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή ΑΘΕΤ. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ ε, επιφυλακτικός ως προς την ευρωπαϊκή πορεία ανάπτυξης και την συμβατότητά της με την Ευρασιατική Ένωση. Ε, το είδαμε ότι δεν μπορούμε να άρουμε τους δασμούς εξαιτίας αυτής της Ένωσης. Αυτό δυσκολεύει τη συνεργασία μας και τις δυνατότητες για τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Αρμενία. Είναι και παραμένει ένα θέμα ε, ενώ στην Ευρασιατική Ένωση ε, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και η κυριαρχία μιας μεγάλης χώρας από την Ένωση αυτή θα πρετανεύουν. Στην Αρμενία όμως είναι και το θέμα του Νοτιού Κάφκασου. Πρέπει να δούμε τη γεωγραφική αυτή ζώνη συνολικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκφραστεί η αλληλεγγύη και η συνεργασία μας προς την χώρα και το λαό της Αρμενίας. Ευχαριστούμε κύριε Οστρεβίτσιους. Ο κύριος Λοντεβίν, ε, Διευθυντής για την Ανατολική Γειτονία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Πρέσβη Μαρκαριάν, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί δίνετε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να πάρει το λόγο ενώπιον της Επιτροπής σας. Στο ανώτατο δυνατό στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο έχουμε παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Αρμενία σε συμφωνία με το Σύνταγμα της χώρας, τις εξελίξεις που έχουν διενεργηθεί και μάλιστα ειρηνικά. Και πρέπει αυτό να το υπογραμμίζω γιατί δυστυχώς δεν ήταν αυτό πάντοτε ε, αυτό που συνέβαινε σε αυτή τη χώρα. Επομένως καλωσορίζουμε ε, τον αυτοπεριορισμό και την αυτοσυγκράτηση και την υπευθυνότητα που έδειξαν όλα τα μέρη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αρμενίας και ε, πιο συγκεκριμένα, όπως ήδη αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες, μέσω της εφαρμογής της Συνολικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε την ομόφωνη στήριξή μας στο Αρμενικό ε, Κοινοβούλιο και υπάρχει σχεδόν ομόφωνη στήριξη ε, και στη δική σας Επιτροπή ε, για τα θέματα αυτά. Ε, αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει την παγίωση της δημοκρατίας στη χώρα αυτή, θα ενισχύσει το κράτος δικαίου, θα, προστατεύσει τα, θα προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα δημιουργήσει μια οικονομία ευημερούσα που θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών της χώρας αυτής. Για να πετύχουμε αυτούς τους σημαντικούς στόχους είναι σημαντικό να γίνεται συνολικός διάλογος μεταξύ όλων των πολιτικών φορέων και εμπλεκομένων φορέων στην Αρμενία. Θα έχουμε προσωρινή εφαρμογή κατά πάσα πιθανότητα από τον επόμενο μήνα και μετά και ε, τότε η φυστάμενη εταιρική σχέση θα γίνει πραγματική συνεργασία και χαιρόμαστε διότι θα συνέλθει το πρώτο Συμβούλιο Εταιρική Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας στα τέλη Ιουνίου, 20 Ιουνίου και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε από δική μας πλευράς. Επίσης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί τα αρμενικά υπουργεία, οι αρμόδιοι και εκπρόσωποι τους ε, συζητούν ήδη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών. Πρόσφατα η Αρμενία υιοθέτησε ένα νόμο ενάντια στην οικογενειακή βία και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ελπίζουμε ότι αυτή η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων και νομοθεσιών θα ευνοήσει το επιχειρηματικό κλίμα και αυτό χρειάζεται γιατί υπάρχουν οι υφιστάμενες ολιγαρχικές δομές πράγματι που ε, πλήττουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τέλος, μας ενδιαφέρουν οι θετικές εξελίξεις και δεσμεύσεις της Αρμενίας στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης και θέλουμε να προωθήσουμε τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ευμερία στην Αρμενία και στην ευρύτερη περιοχή και με χαρά θα καλωσορίσουμε τον Πρωθυπουργό ε, όταν θα ε, κάνει επίσημη επίσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε εδώ. Ε, κύριε Μαρκαριάν, θέλετε κάποια καταληκτικά συμπεράσματα να μας παρουσιάσετε. Εφόσον ναι, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους τους ευρωβουλευτές για τις παρατηρήσεις τους και την διάθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί μας. Φυσικά, θα μεταφέρουμε όλα τα μηνύματά σας. Όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις σχετικά με τις έρευνες ε, καθώς και το εκλογικό δικαστήριο, θα ήθελα να σας πω ότι μόλις τώρα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και μάλιστα όχι επίσημα εντός του Κοινοβουλίου. Εν ευθέτω χρόνο θα σας ε, μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή τύχη στην Αρμενία και έτσι ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Προχωράμε τώρα κατευθείαν σε κοινή συζήτηση για τα θέματα 13 και 14, Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράκ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι τι 12. Μέχρι τις 12 ακριβώς ε, έχουμε διερμηνία, διότι ξεκινήσαμε στις 8 σήμερα το πρωί με την ε, συνεδρίαση του Προεδρείου. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι να περιοριστείτε στο χρόνο σας και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Έχουμε λοιπόν ε, την ε, δεύτερη εξέταση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ. Έχουμε λάβει 138 τροπολογίες και ξέρω ότι η κυρία Σαΐφη εκπονεί προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών. Η κυρία Σαΐφη είναι παρούσα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ελπίζω όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, να αποχωρήσουν σύντομα από την αίθουσα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τις εκλογές που έλαβαν χώρα στο Ιράκ το περασμένο Σάββατο, η ανταλλαγή απόψεων σήμερα μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε εκ νέου τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει έναντι των Ιρακινών προκειμένου να σχηματιστεί και η κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν και προκειμένου να προωθήσουμε έτσι περαιτέρω τη συνεργασία μας για την ανασυγκρότηση, τη συμφιλίωση και τη σταθεροποίηση της χώρας. 138 τροπολογίες έχουν υποβληθεί σε αυτό το σχέδιο έκθεσης και, συμφω... και ευχαριστώ όλους τους κοιόδης εισηγητές και όλους τους βουλευτές για τη συνεισφορά τους. Αυτή τη στιγμή διατυπώνουμε ένα σχέδιο συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχω την αίσθηση ότι πολλές τροπολογίες συμπληρώνουν και λειτουργούν επικοδομητικά ως προς το αρχικό κείμενο. Κάποιες τροπολογίες επιμένουν ε, διότι είναι ανάγκη να μην παραμείνουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα του ΝΤΑΕΣ, του Ισλαμικού κράτους και να βρεθεί τρόπος να ε, προστατευτεί η ποικιλομορφία και ε, η διαφορετική πολιτισμή εντός της Ιρακινής κοινωνίας. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά, να είναι μια κοινωνία πιο συμπεριληπτική που να περιλαμβάνει περισσότερο και περισσότερους μια δημοκρατία σταθερή και ευημερούσα. Αυτά πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών που αποτελούν μέρος των συμβιβαστικών τροπολογιών και θέλουμε ένα κείμενο τελικά που να απεικονίζει τη συνολική κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή στο Ιράκ αλλά να δίνει και όραμα να είναι φιλόδοξο. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον τη συμβολή των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Κύριε Νάρτ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Τόκια, για τη δουλειά σας. Κάνατε εξαιρετική δουλειά και εσείς και τα λοιπά μέλη της ομάδας που και εμείς προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση αυτού του ψηφίσματος. Όπως συνηθίζεται, Ξέρετε, οι καταστροφές που έγιναν με την πολιτικός αναλφάβητη παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών δημιουργούν προβλήματα τα οποία εμείς πρέπει να τα επιλύσουμε. Αλλά και οι Βορειοαμερικανοί επίσης. Στο Ιράκ υπάρχει ένα τεράστιο κενό, ένα τεράστιο χάσμα που θα πρέπει να το καλύψει η ίδια η Ιρακινή κοινωνία. Έχουμε την τύχη να έχουμε τον Αλή Στάνη, ένα θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος ε, ε, έχει μια αντίληψη για ένα Ιράκ που θα περιλαμβάνει όλους. Την καταστροφή αυτή μπορούν να τη λύσουν οι Ιρακινοί χωρίς εκταριστικές αντιλήψεις. Και ε, σε αυτή τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράκ, αυτή η γραμμή είναι που πρέπει να επικρατήσει. Πρέπει δηλαδή το Ιράκ να στραφεί προς τη συμπερίληψη όλων και προς το να ενσωματώσει την πολιτική στην κοινωνία, η οποία ήταν απαραίτητη ε, ως μαχητές για να ε, καταπολεμήσει τους Ισλαμιστές, αλλά τώρα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα και να είναι όλοι μέλος της ίδιας κοινωνίας. Υπήρχε και το θέμα με τους Κούρδους που υπήρξε ο κίνδυνος να ε, κατακαιρματιστεί γεωγραφικά η χώρα του Ιράκ, τα σύνορα και πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να μην έχουμε σεκταριστικές και ιδεολογικές διαιρέσεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και για το Ιράκ και για τις γειτονικέ χώρες. Είναι μια χώρα ε, εξαιρετικά σημαντική σε πολύ εύθραυστη κατάσταση όπου τα, το σημείο ισορροπίας είναι εξαιρετικά λεπτό. Πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Νάρτ. Ε, ε, αν δεν θέλει κανείς άλλος να συμμετάσχει στη συζήτηση, να σας θυμίσω ότι στις 20 Ιουνίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο ή τον Σεπτέμβριο. Θα το δούμε αυτό. Κυρία Σαΐφη, σας ευχαριστώ πολύ για την πολλή δουλειά που έχετε κάνει. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους σκιώδη εισηγητές. Και περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο και τις συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία σας. Δύσκολη η δουλειά μας, δύσκολο το έργο μας. Στις 2.30 θα συνεχίσουμε με, άλλο, με το επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης.